Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, chers collègues, please take your seat. Ich darf alle... Καθίστε συνάδελφοι. Καλώς ορίσατε όλοι σας. Την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών εδώ στις Βρυξέλλες για το τρέχον έτος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών δεν μπορεί να παραστεί σήμερα, γι' αυτό λοιπόν θα προεδρεύσω εγώ. Αλλά έχει και μια ανακοίνωση στις 2 Δεκεμβρίου και στις 17 Δεκεμβρίου δεν πρόκειται να λάβει χώρα η συνεδρίαση τη Επιτροπή Προπολογισμών. Γι' αυτό λοιπόν και σα καλωσόρισα εδώ στι Βρυξέλλε στην τελευταία συνεδρίαση για φέτο τη Επιτροπή Προπολογισμών. Σε περίπτωση που παραστεί κάποια ανάγκη, ενδεχομένω στι 9 Δεκεμβρίου να συνεδριάσουμε στα πλαίσια της Επιτροπής στο Στρασβούργο. Μόνο όμως αν υπάρχει κάποια κατεπίγουσα ανάγκη. Ιδάλλως θα είναι η τελευταία αυτή η συνεδρίαση για φέτος. Η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Όλα λοιπόν ε, όσα ανακοινώνονται και συζητιούνται εδώ πέρα μπορεί να τα ακούσει όλος ο κόσμος. Τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία για την εφαρμογή μπορείτε να τα πάρετε αν θέλετε, αν και νομίζω ότι πιο πολλοί από τους συναδέλφους χαίρονται που την τελευταία εβδομάδα και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον προπολογισμό τον αποφασίσαμε, τον εγκρίναμε στην Ολομέλεια. Äh, δεν είμαι σίγουρη. Άκουσα όμως ότι μια ομάδα Πολωνών δημοσιογράφων πρόκειται να επισκεφτεί την Επιτροπή μας, καλεσμένη του κ. Κοσλόφσκι. Δεν ξέρω αν έχουν καταφτάσει. Να τους καλωσορίσω, αν είναι εδώ. Αχ, εσείς οι δύο είσαστε. Α, μάλιστα. Αυτά παθαίνουμε. Αν φοράμε παροπίδε και δεν βλέπουμε μπροστά στα μάτια μα. Είστε εδώ λοιπόν και οι δύο. Καλώ ήλθατε. Και μα ε, μαγνητοσκοπείτε. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης 17 Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου. Η συνήθι διαδικασία θα ακολουθηθεί. Αν κανείς δεν έχει να κάνει παρατήρηση μέχρι τα τέλη της συνεδρίασης θα, θεωρηθεί, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Τα πρακτικά της 14ης Νοεμβρίου δεν τα έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, αλλά θα τα λάβουμε συντόμως. Όπως θα είδατε, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Ελπίζω όλοι να έχετε τις ε, κάρτες μαζί σας για την ψηφοφορία. Ένας μόνο μου είπε ότι δεν την έχει. Δεν είμαστε όμως και τόσο πολύ Έχουμε οπτική επαφή, αν κάποιος έχει ξεχάσει την κάρτα του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, με τις ψηφοφορίες. So, ähm, Tagespunkt Nummer 8. Στο σημείο 8 λοιπόν της ημερήσιας διάταξης πάμε. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην ε, Παγκοσμιοποίηση Βέστας από την Δανία. Έκθεση του Γιάνν Κοσλόψκη. Να ψηφίσουμε. Εννέα τροπολογίες. Οι πρώτες πέντε τροπολογίες μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Όλοι από την ΕΜΠΛ, Επιτροπή Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνονται λοιπόν. Τροπολογία 6 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Δεύτερο χωρί Δεύτερος κάρτα, μάλιστα, το σημειώνουμε. Ψηφίσατε λοιπόν όλοι. 14 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. Βάιλο και Ρίτσαρντ. Είσαστε υπέρ ή κατά. Υπέρ. Κατά. Κατά κατά λέει η κατα υπερ κατα κατα κατα λεει ο προεδρος Το ξέρω, το ξέρω ότι είσαστε κατά της τροπολογίας αυτής. Τροπολογία 7 και 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Τροπολογία 9 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα, η ηλεκτρονικά, ας ψηφίσουμε επί του συνόλου της έκθεσης. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πολύ ωραία. 24 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια Γιάννου. Το επόμενο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, πάλι για την Νόκια από τη Φιλανδία, αυτή τη φορά. Ο Φαν Ναράνκο Εσκομπάρ είναι ο εισηγητής. Επτά νοητροπολογίες της Επιτροπής Απασχόλησης να ψηφίσουμε από κοινού. Όχι. ποιες δεν θέλετε να συμπεριληφθούν, οι τρία, μάλιστα. Ας τις ψηφίσουμε όλες ξεχωριστά. Ένα, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η τρία. Υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. Η τέσσερα, υπέρ. Η τέσσερα, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η πέντε, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η έξι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 7 υπέρ. Αποχές. Και ποιος είναι κατά, λέει ο πρόεδρος. εγκρίνεται η οκτώ υπέρ. Υπέρ λέω. Η οκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Λείπει μία ψήφος. Όχι, εντάξει. 25 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Να περνάμε στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης First Solar, ηλιακά πάνελα από τη Γερμανία. Τροπολογίες και πάλι από, από την Επιτροπή Απασχόλησης. Πέντε. Να τις ψηφίσουμε από κοινού. Όχι. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Okay. Moment. Inge muss noch okay, ähm, ihre Karte einstecken, ja. 24, 25, no, it's too late. 25, 26. 26 and 3 against. Ja. 26 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. Εγκρίνεται. Και περνάμε λοιπόν. Στα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Αίντερ Ρούμπιαλ. Τρεις τροπολογίες έχουμε της εισηγήτριας. Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού. Η Αίνταρ έχει να κάνει δύο σχόλια από αυτό. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που λαμβάνω το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Υπάρχουν όμως δύο προβλήματα με τις τροπολογίες. Η τροπολογία 5 που εγώ ως εισηγήτρια υπέβαλα στην έκθεση γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα σύνταξης ή μετάφρασης. Νόμιζα ότι στα αγγλικά ήταν αρκετά σαφής, αλλά σε άλλες γλώσσες γίνονται παρερμηνίες. Γι' αυτό προτείνω μία προφορική τροπολογία στη δική μου. Ορίζεται σε ένα κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα υπό τον όρο ότι το εν λόγω κράτος μέλος ή, ή τρίτη χώρα ε, δηλαδή μιλάμε για ένα κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Να καταστεί σαφές. Ε, το δεύτερο θέμα αφορά την τροπολογία Σιλβέστρης όπου συμβαίνει το ίδιο. Ε, διάβασα την τροπολογία στα Ιταλικά και νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα μετάφρασης από τα Αγγλικά στα Ιταλικά η ήρθα σε επαφή μαζί του για να δω κατά πόσο μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά επειδή δεν έλαβα απάντηση, προτείνω να καταψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Είναι ένα θέμα ουσίας, γι' αυτό εάν θέλετε να την υποβάλετε στην αρμόδια επιτροπή θα ήταν σκοπιμότερα. Δηλαδή, προτείνω να καταψηφίσουμε την 11, έτσι ε, ώστε να μην ανακύψουν νέα προβλήματα. Μπορούμε να συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Okay, ε, Μάλιστα. Με τις εξηγήσει και την προφορική τροπολογία, λοιπόν, στην τροπολογία υπαριθμό 5, να ψηφίσουμε την 4 και την 5 και την 6 από κοινού της συγγετρίας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Και περνάμε στις δύο τροπολογίες του Ντομινίκ Ρικέ, 15 και 16. Να τις ψηφίσουμε μαζί. Όχι. Η 15 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η 16 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η τροπολογία 7 και 8 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνονται. Και τώρα περνάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Η 9, Dominique Ρικέ, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 11. Σιλβέστρης. Συμφωνήσαμε να την απορρίψουμε. Υπέρ. Κατά. Κατά. Πολύ ωραία. Και υπέρ, λέει η πρόεδρος. Αποχές. Απορρίπτεται. Σας μπέρδεψα λίγο μάλλον, λέει η πρόεδρος. Περνάμε τώρα σε άλλες τρεις τροπολογίες. Ντομινίκ Ρικέ. Να τις ψηφίσουμε από κοινού. Πολύ ωραία. Η 12, 13, 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άλλες τρεις της εισηγήτριας. 1, 2 και 3. Από κοινού παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. That's it. That's it. Four, four, and two. No, she has the card already. Mm -hmm. has the card. So it's only on mm -hmm. Okay. Haben alle abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. 27 ψηφί υπέρ, μία κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια. Κανονικά θα έπρεπε να ψηφίσουμε για την ανανέωση της Συμφωνίας Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Θα μπορούσαμε να παρακαλέσουμε τους, τον εκπρόσωπο του EFD να πάρει το λόγο, γιατί δεν έχουμε τα έγγραφα στη διάθεσή μας και πώς θα ψηφίσουμε. Εκπροσωπώ τον κύριο Ρολάντα Πάξη, τον συνάδελφο. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για το θέμα. Ευχαριστώ καταρχήν την γραμματεία της Επιτροπής μας για την συνεργασία και υποστήριξη στην σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης. Ελήφθησαν υπόψη οι συστάσεις εμπειρογνωμόνων ένθεν κακήθεν. Θεωρούμε ότι η παράταση, η ανανέωση της συμφωνίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω εμβάθυνση της εργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. προγράμματα που αφορούν την επιστήμη και την τεχνολογία, προάγουν την γνώση και την τεχνογνωσία κατέρωθεν. Η συμφωνία θα βοηθήσει στην διάδοση νέων γνώσεων και θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε νέες αγορές. Στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας θα αφαιρεθούν περίπου 0,55 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι να δώσουμε την δυνατότητα σε επιστήμονες και ερευνητές να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα και να μην ε, περιοριστούν στον ρόλο του συντονιστή. Καλό λοιπόν την Επιτροπή μας να παρακολουθήσει από κοντά την υλοποίηση της συμφωνίας. Η Επιτροπή μας θα υποστηρίξει βεβαίω την ανανέωση της συμφωνίας στον τομέα της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως το 2019. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα υποστηρίξετε την πρότασή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα αν είμαστε υπέρ της ανανέωσης της συμφωνίας ή κατά. Ποιος είναι υπέρ της ανανέωσης της συμφωνίας συνεργασίας, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Κανείς. Εγκρίνεται λοιπόν η ανανέωση. Και τώρα περνάμε στις μεταφορές. Στο συντονιστή του ΕΛΚ να ζητήσω να μας πει κατά πόσον μπορεί να αναλάβει το ρόλο του Τζεβάνι Λαβία. Okay. Eh, Ευχαριστώ. Δυστυχώς ο κύριος Λαβία δεν είναι παρόν σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Ιταλία σήμερα, κάποιο πολιτικό συμβάν ή κάτι που δεν γνωρίζω για τις μεταφορές αυτές, δηλαδή 28, 31 και 32, αυτές οι τροπολογίες σχετίζονται με το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και η θέση του, του εισηγητή είναι ότι θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε αν μπλοκ, διότι ο εισηγητής είναι θετικά διακείμενος. Μετά η 33, η μεταφορά 33, για την έγκριση ε, ενός ε, ειδικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση ε, κινδύνων για τις ΜΜΕ, για την ανάπτυξη και καινοτομία. Η 34 αφορά νέα κατανομή μεταξύ γραμμών ως προς ε, γεωργικά, γεωργικές βοήθειες στο Μαυροβούνιο. Υπάρχουν όμως διοικητικές ελλείψεις και αυτό το είδαμε και σε μία άλλη μεταφορά για τη Φύρομ πρόσφατα. Η θέση του είναι θετική. Η 36 που αφορά 8 εκατομμύρια ευρώ αφορούν αντιμετώπιση ε, καταστάσεων, ε, επιγουσών καταστάσεων. Η 38 είναι μία μεταφορά 70 και 68 εκατομμύριων ευρώ αντιστοίχως από το θεματικό πληρωμών για διεθνείς συμφωνίες αλίες που χρειάζονται για την αλλιευτική συμφωνία με τη Μαυριτανία. Η 40 αφορά μισό εκατομμύριο ευρώ προς διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς για τη διαχείριση αλλιευτικών πόρων. Η 41 παντού υπάρχει θετική γνώμη. Η 41 αφορά ε, τη μεταφορά 300.000 ευρώ για διεθνείς αλλιευτικές συμφωνίες για το ε, πράσινο ακροτήριο και το Κυριμπάτι. Ο εισηγητής, ο Τζοβάνι Λαβία, συμφωνεί και ζητά θετική ψήφο. Επίσης ζητά συγγνώμη για την απουσία του. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση θα ψηφίσουμε όλες τις αιτήσει μεταφοράς ε, τη μία μετά την άλλη. 28, 31 και 32, όντως, καλό θα είναι να ψηφίσουμε από κοινού γιατί αφορούν το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Υπέρ της ε, μεταφοράς 28, ε, 31 και 32. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Να ψηφίσουμε τώρα την 33. Μεταφορά 33. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34. Μεταφορά 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μεταφορά 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Ωραία. Και περνάμε τώρα στα άλλα τμήματα. Προτού όμως ε, ξεκινήσουμε και ακούσουμε τις δηλώσεις του συγκεκριτή, ο οποίος επίσης δεν μπορεί να παραβρεθεί εδώ σήμερα, θα ακούσουμε λοιπόν τον συντονιστή των σοσιαλδημοκρατών. Έχω το καθήκον. Πού είναι ο Γενικός Διευθυντής όμως? Θα πρέπει να ρωτήσω τον Γενικό Διευθυντή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικά κατά πόσον μπορούν να μας μιλήσουν για τις συνέπειες. του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τη μη προσαρμογή των μισθών το 2011. Oui, merci. Euh. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Η Κομισιόν σημείωσε την απόφαση του δικαστήριου. Η απόφαση αφορά ένα διαδικαστικό ζήτημα. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή εξετάζει την απάντηση που, που είναι πιο κατάλληλη ως απάντηση σε αυτήν την απόφαση του δικαστηρίου. Αυτά προς το παρόν και μόνο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Η εξέταση θα συνεχιστεί σε κάθε περίπτωση μέχρι και το επόμενο έτος. Σας είπα ότι σήμερα λαμβάνει χώρα η δική μας τελευταία συνεδρίαση φέτος, εκτός κι αν προκύψει οτιδήποτε έκτακτο, οπότε και θα συναντηθούμε στις 9 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Γι' αυτό λοιπόν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε τα αποτελέσματα της ερευνάς σας από το νέο έτος. Η Μόνικα Χολμάιερ, κοιτάξτε, τα πράγματα τα συγκεκριμένα, τα σημερινά δεν επηρεάζονται γιατί δεν μιλάμε για μεταφορά για το 2011, αλλά έχουμε τη συμφωνία με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που θα υπήρχαν αλλαγές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σήμερα, θα αντιτυπωθεί ένας ε, εκ των υστέρων προποϋπολογισμός σε περίπτωση που προκύψει κάτι από τη δικαστική απόφαση. Αυτό είναι το μοναδικό σαφές. Κατά τα άλλα θα πρέπει να περιμένουμε σε ό,τι αφορά την ε, δικαστική απόφαση η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. <clears throat> Μάλιστα, κοιτάξτε, δεν θα επισέλθουμε όμως στην, ε, στις λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη δικαστική απόφαση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Τώρα, να ακούσουμε τον Ιβάιλο από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ο κύριος Ορτού. Mm ο κ. Χάρτον, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή σημείωση σε ό,τι αφορά το C8. Σε ό,τι αφορά την αγορά iPads, ε, ταμπλέτες ε, γενικά. 1.100 ταμπλέτες με, ε, με μία σύμβαση με μια σύμβαση εξυπηρέτηση. 1.363 ε, ευρώ δηλαδή για κάθε ταμπλέτα. Μου φαίνεται είναι πάρα πολύ ακριβό. Τι να σα πω. Wir fragen ähm, θα ζητήσουμε την, ε, να μας απαντήσει η γραμματεία, αλλά να μας μιλήσει η Ingeborg καταρχάς. καταρχάς. Να σας υπενθυμίσω τι θα γίνει ε, με τα χρήματα τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν. Να σκεφτούμε δηλαδή και το ποσό το οποίο δεν αξιοποιείται. Για τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό με ενδιαφέρει, λέει η κυρία Γκρέσλε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μία νέα πρόταση και δεν ξέρουμε τι ποσό θα μείνει αχρησιμοποιητό γιατί δεν έχουμε εξαγάγει τα θετικά συμπεράσματα. Αν σωστά κατάλαβα τον κύριο Γενικό Διευθυντή, μας ανέφερε ότι αυτό που αποφάσισε το δικαστήριο είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία Δηλαδή, δεν αποφάνθηκε καν για το ύψος της προσαρμογής των μισθών. Καταρχάς αποφάνθηκε για την διαδικασία, το ποιες θα είναι οι συνέπειες. Αυτό θα μας το πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου. Και ενδεχομένω να καταρτιστεί ένα εκ των υστέρων προπολογισμό. Άρα για το ποσό δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι στην παρούσα φάση. Η κυρία Γκρέσλε, κοιτάξτε. Το ερώτημα ήταν, είναι τι προπολογισμό ε, προβλέπεται για αύξηση των μισθών. Και η διαδικασία του δικαστηρίου λέει ότι... Α, δεν λέει τίποτα. Η Ευρωπαϊκή, ε, το Ευρωπαϊκό το δικαστηρίο λέει ότι μπορεί να κάνει μία πρόταση καινούργια και η άρνηση του Συμβουλίου είναι εντάξει. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσο θα κάνει νέα πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Μπορούμε να το ερμηνεύσουμε λοιπόν είτε έτσι είτε αλλιώς. Καλό θα ήταν λοιπόν να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα το χειριστεί. Αλλά είναι πολιτικό το θέμα. Η κυρία Πρόεδρος, κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποιο αριθμητικό στοιχείο, όμως δεν έχουμε αποφασίσει κάτι στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό λέγαμε όλη την ώρα, ότι δεν είναι αυτός τρόπος να κάνουμε προπολογισμό. Και αυτό λέγαμε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ασκεί πίεση στο Συμβούλιο. Δεν ξέρουμε όμω τελικά τι γίνεται, γιατί πολύ απλά δεν περιλαμβάνει τίποτα. Δεν αποφάσισαμε τίποτα στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται. Τα μέτρα με τα οποία προσπαθούμε να ασκήσουμε ε, επιρροή και πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει τον ε, προπολογισμό όπως πρέπει, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ε, μέσα πλέον, να βαριέται και ο Ιβάιλο για, μίλα μας Ιβάιλο, για τις μεταφορές στους άλλους, στα άλλα τμήματα. Nobody can be... Κυρία Πρόεδρε, κανείς δεν πλήττει εδώ. Πριν μιλήσουμε για τις προτάσεις μεταφοράς κονδυλίων να προσθέσω μια πρόταση στην προηγούμενη συζήτηση. Όταν κρίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι απάντηση θα δώσει, θα ασχοληθούμε και εμείς με το θέμα. Αλλά είμαστε έτοιμοι εν ώψη του πολιτούς δημοσιονομικού πλησίου. Τώρα, όσον αφορά το... Ε, και εξονόματος του τέρκβον, ο οποίος ε, δυστυχώς ε, δεν μπορούσε να έρθει στη Βρυξέλλη σήμερα λόγω άλλη υποχρέωση. Θα ήθελα να προτείνω διάφορες μεταφορές. Οι περισσότερε αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον προπολογισμό του. Πρόκειται για μεταφορές που αφορούν την ενίσχυση του Ταμείου για, το, την εκδήλωση την Ευρωπαϊκή Νολέα του χρόνου, European Youth Event, επίσης για εξοπλισμό πληροφορικής, για το σύστημα CISPER συγκεκριμένα και για επιπλέον εξοπλισμό για συσκευέ που χρειαζόμαστε συγκεκριμένα. Και μετά το 9 αφορά πληρωμές για τα πάνε ταξιδίου των βουλευτών. Επισημένω το γεγονός ότι ίσως πρέπει να βραχυνθεί η περίοδος των δύο των εντός των οποίων μπορεί να υποβληθεί αίτηση αποζημίωσης για έξοδο ταξιδίου. Πολλά τα δύο χρόνια. Μετά έχουμε κάποιες μεταφορές που αφορούν, που αφορούν τους μισθούς των βοηθών των βουλευτών και μετά προκαταβολές για το κτίριο στο Λουξεμβούργο που έχουν ζευτεί από 85 διαφορετικές ε, γραμμές. Υποτίθεται ότι μας εξοικονομεί κάποιους τόκους αυτή η υπόθεση επιτρέπονται αυτές και προτείνονται οι εν λόγω μεταφορές. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να σχολιάσω και τις άλλες μεταφορές που προτείνονται προκειμένου σε αυτή τη φάση, αφορούν την εποπτική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε μόνο για 80.000. Πρόκειται για εσωτερική μεταφορά από τη Διερμηνία σε έξοδα κτηρίου. Είμαι υπέρ αυτών των μεταφορών ως εισηγητής και τις ε, προτείνω. Μάλιστα, πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, να σας παρακαλέσω να απαντήσετε σε ό,τι αφορά το ερώτημα για την τιμή για τις ταμπλέτες. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως το βλέπετε και στο προτείνωμενο κείμενο για τις μεταφορές, το μέσο εκτιμωμένο κόστος της, του κάθε είναι 854, 854 συμπεριλαμβάνονται όμως και υπηρεσίες που αφορούν την υποστήριξη, το help desk, συντήρηση και εγκατάσταση συγκεκριμένων εφαρμογών που είναι απαραίτητες για τους χρήστες στο πλαίσιο του e-committee, e-meeting κλπ. Αυτό θα εξοικονομήσει χαρτί θα μειώσει τον αντικτυπώμα μας στο περιβάλλον λόγω διοξιδίου του άνθρακα. Οι συσκευέ αυτές θα πάνε κυρίως στα χέρια υπαλλήλων στο Squared Maze και θα βελτιώσει την παραγωγικότητά τους μέσω ακριβώ της χρήσης ε, αυτών των νέων τεχνολογιών. Επίσης, τον Ιούνιο του 2014 θα εφοδιαστούν και οι βουλευτές με δοκιμασμένες εφαρμογές για τον ίδιο σκοπό για να μην χάσουμε μήνες μετά από τις επόμενες εκλογές. Να έχουμε δηλαδή τα εργαλεία αυτά ήδη στη διάθεσή μας και να είναι και επιχειρησιακά έτοιμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θεωρώ δεδομένο ότι οι βουλευτές στην περίπτωση αυτή θα τα λάβουν τα μηχανήματα αυτά τον Ιούλιο τον νωρίτερο, όταν θα έχουν εκλεγεί και θα έχουν ξεκινήσει εδώ τη νέα θετία. Ήθελα μόνο, κυρία Χολμαϊρ, το θέμα δεν είναι οι βουλευτές, το θέμα είναι ότι αυτά τα μηχανήματα θα τα πάρουν ε, το διοικητικό προσωπικό. Βάλαμε τα έξοδα αυτά στο paperless. Δεν μιλάμε δηλαδή... Ε, δεν μιλάμε μόνο για το πλήρως, δεν είναι μόνο το κόστος που υπάρχει, είναι και η μείωση στον προπολογισμό σε άλλους τομείς. Μάλιστα, να τα ψηφίσουμε όλα μαζί, λέει η Πρόεδρος. Όχι, κάθε αίτηση μεταφοράς ξεχωριστά. Να ξεκινήσουμε στο C4, υπέρ της μεταφοράς. Κατά. Αποχές. Δεν κρίνεται. C7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. C8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. δεν έχουμε μόνο την αίτηση μεταφορά, αλλά και την ομάδα εργασίας μας θα την ε, δώσουμε την εντολή σε ό,τι αφορά το χρονικό διάστημα που γίνεται ο υπολογισμό να μπορεί να συντομευτεί το διάστημα αυτό προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ε, προγραμματισμό. Θεωρώ ότι ένας χρόνος αρκεί, δεν χρειάζεται δύο χρόνια. George, Μόνικα, όποιος θεωρεί ότι πλήττεται, να το θίξει αυτό στην ομάδα εργασίας. Δεν θεωρώ ότι έχει άμεσο αντίκτυπο, αλλά είναι βελτίωση. Αυτό θεωρώ εγώ. Λοιπόν, μαζί με το C9, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. C10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. C12 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και τώρα... Ο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Μάλιστα. Περνάμε τώρα στην εκτηριακή πολιτική. Και σε κάθε περίπτωση σήμερα θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτά που θα μας εξηγήσει η Μόνικα. Στα κτίρια φτάσαμε στην κτηριακή πολιτική. ich darf zunächst einmal ε, eine θα ήθελα καταρχάς να σας απευθύνω μία έκκληση, μία απλή έκκληση. Θα πρέπει τα δύο απλά project για την κτηριακή πολιτική Κόλτπελ στο Λουξεμβούργο Κάπου θα πρέπει να τους βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους που φιλεξινούνται στο κτίριο αυτό. 1,5 εκατομμύρια λοιπόν εξοικομονούμε το ίδιο κτίριο με πιο ευνοϊκούς όρους. Και μας υποσχέθηκαν μάλιστα ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε ε, ανακαίνιση. Βελτιώθηκαν λοιπόν οι όροι. Σαφώς. Ελπίζω να συμφωνήσετε για να μην χρειαστεί να το συζητήσουμε στις 9 του μηνός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από πλευρά των συναδέλφων. Να μην γνωμοδοτήσουμε δηλαδή, απλά να πούμε ότι συμφωνούμε. Μάλιστα. Να το ολοκληρώσουμε. ΕΜΠΑ. Η ΕΜΠΑ είναι λίγο πιο περίπλοκο θέμα. Και γιατί? Γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική δεν έχει καταφέρει να κάνει αναφορές ε, όπως χρειαζόταν. Έχουν κάνει συμβάσεις τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους που από πλευρά Συμβουλίου και Κοινοβουλίου έπρεπε να εγκριθούν. Τα σύνορα, τα όρια τα οποία προβλέπονται στην, ε, στο, ε, στην, στον κανονισμό για τον προϋπολογισμό θεωρώ ότι έχουν ξεπεραστεί. Σαφέστατα, πρώτη φορά λοιπόν παρουσιάζεται τέτοιο φαινόμενο. Μέχρι τότε τσακωνόμασταν, μέχρι σήμερα τσακωνόμασταν για τις τιμές. Και λέγαμε για παράδειγμα στο Λονδίνο ότι ήταν πολύ υψηλέ οι τιμές. Τώρα όμως πραγματικά μιλάμε για σύμβαση μίσθωσης χωρίς έγκριση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Πρώτη φορά. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει καταρχάς να επισημάνουμε αυτή την παραβίαση Κατά δεύτερον, ότι πρόκειται για υπερβολικά υψηλό κόστος, επειδή το κτίριο αυτό είναι πολύ πιο ακριβό από την υπηρεσία την ιατρική, για την οποία τότε διαμαρτυρόμασταν τιμή, μέση τιμή για ένα τραγωνικό μέτρο πάνω από 1000 ευρώ. Είναι πραγματικά εξωφρενικό αυτό που περιλαμβάνεται στη συμφωνία και επιπλέον το κόστος για 1,5 έτος και για τα έπιπλα και για την ε, αλλαγή της διαρρύθμισης είναι πιο υψηλό από το ενίκιο. Έχουμε και τις ε, υπηρεσίες σύμβουλων. Στον ένα το όροφο, για παράδειγμα, είναι ήδη εκμισθωμένο ένα τμήμα και η ιδέα ήταν να εκμισθωθούν και άλλα δύο τμήματα ε, δεν είναι τόσο περίπλοκο σαν ιδέα, γιατί πληρώσαμε 100.000 και παραπάνω σε υπηρεσίες παροχή συμβουλών, δεν ξέρω. Κανονικά η ΕΜΠΑ νομίζω ότι θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να μας έχει υποβάλει αυτά τα σχέδιά της, τα μακροπρόθεσμα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να είμαστε και γρήγοροι. Αλλά τώρα δεν γίνεται να αποφασίζουμε έτσι τελευταία στιγμή. Τώρα λοιπόν έχουμε το εξή πρόβλημα. Αν πούμε ότι θεωρούμε ότι όλο αυτό το οικοδόμημα είναι παράνομο και θα πρέπει να λυθούν αυτές οι συμβάσεις, αυτό θα μας κοστίσει ακόμα πιο πολλά λεφτά. Άρα, εγώ τι προτείνω, να αναφέρουμε ότι είναι παραβίαση του κανονισμού για τον προπολογισμό. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαγάγει τα απαραίτητα συμπεράσματα προκειμένου να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να μην τηρεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ας πούμε, τις ε, προθεσμίες αυτές. Θα πρέπει οι υπηρεσίε αυτές να τηρούν τους κανόνες που προβλέπονται. Και το γεγονός ότι πρόκειται ακριβώς για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας των Τραπεζών με απογοητεύει ε, πολύ. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι άλλωστε και τόσο περίπλοκος ο κανονισμός για τον προϋπολογισμό. Αν θέλουμε λοιπόν, ε, εκεί είναι μπορούμε να τον διαβάζουμε. Νομίζω ότι μια αρχή υποπτία τραπεζών λογικά διαβάζει και πιο ε, και δύσκολους, δύσκολα κείμενα από ότι αυτό. Έπρεπε να έχει τηρήσει τους κανόνες. Το ελεκτικό συνέδριο λοιπόν θέλουμε να ελέγξει τις συμβάσει, να εξετάσει κατά πόσον υπάρχουν και άλλα προβλήματα ενδεχομένω. Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας των Τραπεζών να μην μας αποστείλει ξανά εκ των υστέρων αυτό το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τα κτίρια. Διάλεξα λοιπόν μία διατύπωση που αναφέρει ότι δεν μπορούμε να εγκρίνουμε γιατί δεν προβλέπεται από τον κανονισμό έγκριση εκ των υστέρων, αλλά δεν ζητούμε καταγγελία των συμβάσεων μίσθωσης, γιατί αυτό θα κόστιζε ακόμα πιο πολλά χρήματα και δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να προκαλέσουμε ακόμα μεγαλύτερη ε, πολυπλοκότητα και να παραλύσουμε και την ΕΜΠΑ. Να ζητήσουμε όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να μην συμβεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο και να ελέγξει τον υστέρων τι συνέβη. Ελπίζω οι συνάδελφοι να συμφωνήσουν. Προσπάθησα να μην είμαι πάρα πολύ επιθετική στη διατύπωσή μου που πραγματικά ζορίστηκα πάρα πολύ σε ό,τι αφορά και αυτή τη διατύπωση για τις συμβάσεις ε, εκμίσθωσης και ο Επίτροπος Μπαρνιέ ανέφερε σε μία συζήτηση ότι το θέμα αυτό θα τον απασχολήσει και θα υπάρξουν και συνέπειες σε ό,τι αφορά αυτούς τους εξωτερικούς οργανισμούς προκειμένου να μην μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να σας τα παρουσιάσω και πιο όμορφα από ό,τι είναι. Μάλιστα. Σας καλώ λοιπόν να υπερψηφίσετε και να υποστηρίξετε αυτή την τοποθέτησή μου. Θα τα ακούσουν, λέει η Πρόεδρος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Τζορτζ Λάιεν. Hm? Uh, uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τη Μόνικα, είμαι και εγώ θυμωμένο με αυτό το επεισόδιο. Δύο θέματα έχουμε εδώ. Το ένα είναι η διαδικασία δημοσιότητα. και εδώ υπάρχει μια σειρά αστοχιών στην έκτος όσον αφορά την τήρηση της διαδικασίας. Έχετε δίκιο. Μπορούμε να απορρίψουμε τα πάντα, αλλά αυτό θα κοστίσει περισσότερο. Και ουσιαστικά μας λένε, συμφωνήστε για να μην πληρώσουμε περισσότερα. Είμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος, όπως λέμε. Το θέμα είναι να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Να στείλουμε το μήνυμα λοιπόν το μήνυμα που πρέπει στην ΕΚΤ. Να ξέρουν ότι την επόμενη φορά, αν δεν κάνουν το σωστό, εμείς δεν θα, έχουμε κανένα, δεν θα διστάσουμε καθόλου και θα αναπέμψουμε οποιαδήποτε πρόταση. Ιδιαίτερα μετά από απόφαση δικαστηρίου περί Μετά, η αξία η χρηματική της απόφασης. Και εδώ έχει σπαταληθεί χρήμα. Αυτή είναι η εντύπωσή μα. Εμεί ω ε, βουλευτέ βεβαίω δεν είμαστε και ειδικοί γι' αυτό και επελήφθη το ελεγκτικό συνέδριο. Θέλαμε όμω και εμεί ω Επιτροπή να ρίξουμε μια ματιά. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να τους επιπλήξουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και είμαι σίγουρο ότι η συνάδελφος θα το πράξει. Λοιπόν, δύο είναι τα σημαντικά ελαττώματα. Το ένα είναι της διαδικασία και το άλλο της πραγματική αξία αυτής της σύμβασης. Θα δούμε αυτά όταν μα στείλει την έκθεσή του το ελεγκτικό συνεδρίο, αλλά εν πάση περιπτώσει η Επιτροπή μα πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι την επόμενη φορά οποιαδήποτε αστοχία θα οδηγήσει στην απόρριψη μελλοντικών συμβάσεων. Σα ευχαριστώ πολύ. Ναι, Μόνικα, εσύ θα πάρεις το λόγο πάλι στο τέλος. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στο Γιέντ Γκάιερ, Ντόμινεν Ενρικέ, Ρίτσαρτ Άσχορτ και δεν ξέρω. Να πάρεις το λόγο μετά. Ναι, είπατε κι εσείς σε μια σημαντική λέξη. Ε, πρέπει να το υπενθυμίσουμε, να το αξιολογήσουμε πολιτικά και να θυμίσουμε ότι υπήρξε απόφαση του Συμβουλίου με την οποία οι τρεις αυτές οι οργανώσεις στη Φραγκφούρτη, Παρίσι και στην Φραγκφούρτη, στο Λονδίνο και στο Παρίσι ε, ιδρύθηκαν για διάφορους λόγους. Στην περίπτωση του Λονδίνου το Συμβούλιο αναγκάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να νοικιάζει ένα κτίριο στην πιο ακριβή αγορά ακινήτων του κόσμου και αυτό τη στιγμή που θα μπορούσε αυτό το ακίνητο να το νοικιάζει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος τη Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν ξέρω ποιο είναι ο λόγος γι' αυτό, αλλά να διευκρινίσουμε ποιο φέρει τις ευθύνε, Να διευκρινίσουμε ότι δεν ήταν επιθυμία εδώ του Κοινοβουλίου να γίνει αυτό, να τοποθετηθεί δηλαδή αυτή η υπηρεσία στην πιο ακριβή αγορά κινήτων του κόσμου. Μία ερώτηση προς τη Μόνικα τώρα. Αυτή η διαδικασία εκμίσθωσης καθοδηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, EBA και πώς, ε, ποια είναι η σύνθεση του Συμβουλίου αυτού σε περίπτωση που υπάρχει ήδη κάτι τέτοιο. Όλες τις ερωτήσεις, λέει η Πρόεδρος, θα τις γράψει η Μόνικα, θα τις σημειώσει για να τις απαντήσει στο τέλος. Είμαστε απογοητευμένοι, αλλά σίγουρα έχουμε φυγεί, γιατί τέτοιες δαπάνες και τέτοιο κόστος είναι υπέρογκο, δηλαδή δεν σχετίζεται καν με την αγορά του Παρισιού. Άρα ε, αυτοί που ασχολήθηκαν δεν έδειξαν την κατάλληλη ε, στάση ε, αυτοί που υπογράφουν τις συμβάσεις, ε, ποιον εκπροσωπούν, ποιος τους προσλαμβάνει και πώς μπορούν να μην εφαρμόζουν τον κανονισμό. Όταν μου λέτε ότι αν προσβάλλουμε τις συμβάσεις αυτό θα στοιχήσει ακόμα περισσότερο, θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο αυτός που υπέγραψε ε, είχε τις προϋποθέσεις και τα εχέγγυα να κάνει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι ο διευθυντής του οργανισμού το έκανε. Πώς μπορεί να δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι αυτών των οργανισμών πέρα από τον κανονισμό και χωρίς προγενέστερη αδειοδότηση που να συνάδει με τη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει υπάρχει ε, ένα συμβατικό κύρος, μια συμβατική εγκυρότητα. Εάν είχε το, το κύρος για κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ε, διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, είναι λυπηρό αυτό που γνωρίσαμε και σκανδαλώδες θα μπορούσα να πω, αλλά θα πρέπει να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί, όπως είπε η Μόνικα, και να επιβάλλουμε κυρώσεις τη στιγμή που όλοι φέρουν ευθύνη όταν κινούνται πέρα από την ε, διαδικασία. Ε, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι υπέτοι και να φτάσουμε στις συμβατικές συνέπειες που επιβάλλονται. Σας ευχαριστώ, ο Um, Chairman, thank Συμφωνώ με αυτά που είπε η Μόνικα. Ε, πολύ σωστή η στάση της. Και η όλη κατάσταση είναι απαράδεκτη. Είχαμε ε, πολλές αποτυχίες, δηλαδή δεν ε, ακολουθήσαμε τον κανονισμό που έχει οριστεί και γιατί πρόκειται για μια ενία τραπεζική αρχή που δεν μπορεί να ακολουθήσει τους κανονισμούς. Άρα δεν, ε, έχω, δεν εμπιστεύομαι αυτή την τραπεζική αρχή. Από όσο γνωρίζω, η επιλογή του κτηρίου είναι ακατάλληλη για το έργο τους. Αυτό βεβαίως είναι εκτός ελέγχου του Κοινοβουλίου, αλλά φαίνεται παράλογο το ότι ο οργανισμός της ε, υγείας που βρίσκεται στο Canary Wharf αφορά έναν τομέα ο οποίος ασχολείται με χρηματοοικονομικά όπου θα μπορούσε να ε, έχει την έδρα του σε αυτό το σημείο και όχι στο, και όχι στο City του Λονδίνου. Όταν τους ρώτησα γιατί, μου είπαν ότι βρίσκεται πιο κοντά για λόγους ε, ε, επικοινωνίας και υποδομής, αλλά αυτό δεν με έπεισε. Η Μόνικα προέβαλε μία πολύ λογική λύση. Δεν έχουμε και τόσες επιλογές. Προσβλέποντας το μέλλον, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Πολλοί συνάδελφοι ε, ε, ζήτησαν από το ελεγκτικό συνέδριο να αποφανθεί και συμφωνώ με αυτό. αλλά θα πάρει πολύ καιρό και δεν μπορεί να ισχύσει αναδρομικά. Μέσα στα πλαίσια της ε, Επιτροπής μπορούμε να ζητήσουμε από την ε, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή να έρθει ενώπιόν μας και να μας δώσει εξήγησης. Ναι, ναι, το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Μπορούμε να το ζητήσουμε κατευθείαν, γιατί την πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο όμως ε, έγινα έξαλλη. Και θέσαμε κάποιες ερωτήσεις τότε στον διευθυντή. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Να δώσω το λόγο όμως καταρχάς στον Σαλβαδόρ και στον Γιάννη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομη η ερώτησή μου και πολύ συγκεκριμένη. Σε αυτή την περίπτωση ποιος προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και με ποιο τρόπο. Uh, Ευχαριστώ Παρακολουθώ τη συζήτηση, δεν γνωρίζω την περίπτωση, αλλά η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Μπορεί αυτό να παραμείνει χωρίς συνέπειες, διότι ε, παραβαίνει κανείς τον νόμο και αυτό θα το δεχτούμε, θα λάβουμε γνώση χωρίς να επιβάλλουμε Αγγέλικα. Η Αγγελικά. Ευχαριστώ αν έχουμε δυνατότητα επιβολή κυρώσεων, νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους αυτοί που πρέπει να την αναλάβουν. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα. Πρόεδρος, όχι. Αυτό το ερώτημα δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν και είπε η ότι θα πρέπει να το ζητήσουμε αυτό και από πλευρά Ευρωπαϊκού Ανεκτικού Συνεδρίου και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένω να μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση στην νομική μα υπηρεσία για το θέμα αυτό. Προτού όμω απαντήσει η Μόνικα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Διευθυντή τη EBA, τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Δεν θα μπορέσει να μα δώσει κάποια εξηγήση, αλλά θα μπορούσε να πάρει το λόγο να πει δύο κουβέντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ γιατί με καλέσατε εδώ. Βεβαίω, δεν έχουμε επαρκή χρόνο για να επεξηγήσουμε την όλη διαδικασία στην Επίτροπη Προϋπολογισμών. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι είμαι έτοιμος να έρθω ενώπιον σας λογοδοτώντας και εξιστορώντας τι ακριβώς συνέβη είτε στην Υποεπιτροπή είτε στην Ολομέλεια της Επιτροπής. Ποιος υπέγραψε τη σύμβαση εγώ. Εγώ είμαι ε, εκτελεστικός διευθυντής της ε, αρχής αυτής, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Είμαι ενώπιόν σας λοιπόν. Η αρχή αυτή όταν άρχισε τις δραστηριότητες της το 2011 είχε συμβάσει στο κτίριο που βρίσκεται σήμερα Άρα δεν ήταν επιλογή, δεν ήταν δική μας η επιλογή του κτηρίου. Ε, καταλαμβάναμε ένα μέρος του κτηρίου όπου στεγαζόταν η αρχή, διότι όπως ξέρετε. Ε, στην αρχή είχαμε μία επιτροπή τύπου 3 και ε, είχε συγκεκριμένο νομικό χαρακτήρα. Γι' αυτό στην ουσία κληρονομήσαμε αυτές τις συμβάσεις. Όταν εγώ προσήλθα στην αρχή ήταν μια πολύ μικρή οργάνωση και ήθελε να αυξήσει το προσωπικό και τις δραστηριότητες ε, δυνάμει του κανονισμού για τη συγκρότηση της αρχής. Όταν ανέλαβα εγώ καθήκοντα, Αμέσως αρχίσαμε τη διαδικασία προμηθειών για να βρούμε ένα σύμβουλο ακίνητης περιουσίας, για να βρούμε ε, ε, μία ε, συγκεκριμένη στέγαση στο Λονδίνο. Και αυτό είχε αποφασιστεί όταν εγκρίθηκε ο ιδρυτικός κανονισμός της αρχής. Άρα, συμμορφωθήκαμε απόλυτα με βάση μία σύμβαση που υπογράψαμε στο τέλος του χρόνου. Είχαμε και σύμβουλο ακινήτων, ήταν μία μακρά διαδικασία και υπογράψαμε στα τέλη του 2011. Στη συνέχεια, ήδη είχαμε επεκτείνει τις δραστηριότητές μας αυξήθηκε το δυναμικό της αρχής και τριπλασιάστηκε μέσα σε μία διετία. Μετά, στην αρχή του 12, με τη βοήθεια του Συμβούλου Ακινήτων, κάναμε μία έρευνα της αγοράς. Εξετάσαμε διάφορες, διάφορα σημεία του Λονδίνου, όπως το City και το Canary Wharf, και όπως καταλαβαίνετε, διαφορετικά σημεία δίνουν και ένα σχετικό πλεονέκτημα, σχετικά πλεονέκτηματα. Και θεωρήσαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα μικρό κατάλογο ε, κτηρίων και αποφασίσαμε να μεταφερθούμε το 13 σε ένα άλλο κτίριο, διότι όπως είπε η κυρία ε, Χολμάιρ, στο, στην εκμήθωση που υπήρχε, υπήρχε μία ειδική ρήτρα που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος του 12. Άρα θα, ε, αν, δεν, αν μάλλον καταγγέλαμε αυτή τη σύμβαση, τότε θα έπρεπε να ε, μικρύνει το χρονικό διάστημα μίσθωσης κατά ένα χρόνο. Το ατυχές ε, γεγονός, οι ατυχείς εξελίξεις αποτελούν ένα γεγονός και εδώ δέχομαι τις επικρίσεις σας. Εγώ ήρθα σε επαφή με τον εισηγητή πολύ αργά για την διαδικασία έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό. Και τότε έπρεπε να καταγγείλουμε τη σύμβαση ακολουθήσαμε μία διαδικασία διαγωνισμού, επιλέξαμε ένα κτίριο που ήταν πιο φτηνό και αυτό θα αρκούσε για ε, την αρχή με βάση τις ε, εκτεταμένες της δραστηριότητες. Χάσαμε λοιπόν αυτή την προθεσμία με βάση τη ρήτρα καταγγελίας και παραμείναμε στο ίδιο κτίριο και πρέπει να περιμένουμε τη λήξη της σύμβασης. Εγώ ήρθα σε επαφή με τον ιδιοκτήτη και τον ρώτησαν μπορεί να ε, μειώσει το μίσθωμα φτάνοντας στο επίπεδο του μειοδοτικού διαγωνισμού, δηλαδή ε, να έχουμε τους ίδιους όρους και μειωμένη τιμή, όπως αποφασίστηκε στο μειοδοτικό. Ήρθαμε λοιπόν σε επαφή με την DG Markt με τις οικονομικές αρχές για να ε, έχουμε τη συμβουλή της Επιτροπής και μέχρι το τέλος του 12 με μια επιστολή του Ιανουαρίου του 13 του τρέχοντος έτους ε, μάθαμε ότι θα πρέπει να αρχίσουμε μια νέα διαδικασία επιλογής. Αυτό επιθυμούσε η Δημοσιονομική Αρχή. Στο μεταξύ έπρεπε να επεκτείνουμε ε, το, έπρεπε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες και έπρεπε να βρεθούμε αλλού γιατί έχουμε 59 ε, τεχνικές προδιαγραφές προς την Επιτροπή και είχαμε 60 παρόντες σε πολλές ε, τεχνικές συνεδριάσεις. Δεν είχαμε λοιπόν τους χώρους για να γίνουν αυτές οι δημόσιες ακροάσεις και να ανταποκριθούμε στο έργο μας με συμβούλεψαν τον Ιανουάριο γραπτός να προχωρήσω με την υπογραφή του, της σύμβασης, της βραχυπρόθεσμης σύμβασης και μετά να αρχίσουμε μία πιο μακροχρόνια επιλογή με την διαδικασία που ισχύει, να γίνει δηλαδή μία νέα επιλογή και μία νέα διαδικασία έγκρισης με βάση το δημοσιονομικό κανονισμό. Εγώ υπέγραψα τη σύμβαση το Φεβρουάριο όπως είπε και η κυρία Χολμάιερ και όπως αναφέρεται και στη γνωμοδότηση, δυστυχώς επειδή ε, λόγω μάλλον της ε, βραχυχρόνιας ε, προθεσμίας της σύμβασης και επειδή οι συμβάσεις λήγουν το ίδιο χρονικό διάστημα, αν θέλουμε να μετακινηθούμε μπορούμε να μετακινηθούμε. Άρα υπογράψαμε αυτές τις βραχυχρόνιες συμβάσεις που ισχύουν για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Άρα το μίστομα είναι υψηλό. Ε, η διαδικασία έρευνας της αγοράς βασίστηκε σε διαγωνισμούς. Πάντα χρησιμοποιήσαμε τη διαδικασία μειοδοτικού ε, διαγωνισμού τα έπιπλά μας ε, έχουν αγοραστεί από δεύτερο χέρι, άρα δεν κινηθήκαμε καθόλου εκτός κανονισμού κατά την αγορά κατά τις αγορές που έπρεπε να γίνουν, που εντάξει κατανοώ ότι είναι ακριβές. Έχουμε λοιπόν αυτές τις, ε, ισχύει αυτή η σύμβαση μέχρι του χρόνου Έχουμε αρχίσει την διαδικασία μακροχρόνιας επιλογής με ρήτρα καταγγελίας. Στείλαμε τα σχετικά έγγραφα στη Δημοσιονομική Αρχή, το Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και είμαστε στην τελική φάση επιλογής με την DG έτσι ώστε να προχωρήσουμε με την πλήρη έγκριση της διαδικασίας επιλογής. Αυτή είναι μια σύνοψη του τι συνέβη και θα ήθελα να πω ότι αυτά ήταν τα κίνητρά μας, μάλλον η διαδικασία, γι' αυτό ακολουθήσαμε αυτή τη διαδικασία και είμαι έτοιμος να προσέλθω ενώπιον σας οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για όσο χρειαστεί για να σας επεξηγήσω ε, σαφώς τι έγινε με λεπτομέρεια. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μακρηγορήσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξηγήσει που μα δώσατε. Η Μόνικα Χόλμα έχει το λόγο. Μη με παρεξηγήσετε, αλλά να βάλω λίγο νερό στο κρασί σας. Καταρχάς, ε, δεν κοστίζουν λιγότερα τα τετραγωνικά μέτρα. Δεν ε, ε μισθώσαμε πιο μικρή επιφάνεια. είναι σαν να μου πείτε ότι, κοιτάξτε, ε, έχουμε ένα ωραίο σπίτι, καλή τιμή ένα τετραγωνικό, αλλά θα πρέπει να πληρώσουμε την ανακαίνιση. Όχι, μέχρι 1300 ευρώ αν τετραγωνικό μέτρο έχουμε φτάσει τιμή, σε τιμές. Ακόμα και για το μέρος αυτό στο Λονδίνο είναι πολύ υψηλό το κόστος. 195.000 έχουμε έξοδα δαπάνες για consulting, έχουν υπογραφεί αυτές οι συμβάσεις και δεν μπορούν να ακυρωθούν, δεν μπορούν να καταγγελθούν. Τον Μάιο του 2012, όταν κάναμε την πρώτη συζήτηση, κάναμε διάφορες τηλεφωνικές συνομιλίες με το γραφείο και με τους αρμόδιους ε, υπαλλήλους και τον, με τον κύριο Παλκασέψ μιλήσαμε, όπου όχι μόνο υπέδειξα ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη κοινοποίησης, αλλά επέμεινα και σε αυτή. Είπα το συντομότερο δυνατόν να μας στείλουν τα στοιχεία αυτά. Επίσης, ε, στείλαμε στον ε, διευθυντή τα σχετικά, τα σχετικά προβλήματα, τα επισημάναμε. Το θέμα λοιπόν δεν ήταν μόνο τέλη Ιουλίου, μάλλον υπήρχε ένα λάθος στην ημερομηνία, ε, τέλη Ιουλίου και όχι τέλη Ιουνίου. Θα μπορούσαμε να έχουμε κινηθεί πιο γρήγορα και να είχαμε δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε ό,τι αφορά αυτή την οργάνωση, αυτή την εξωτερική υπηρεσία. Αυτό τώρα που αναφέρω στη γνωμοδότησή μου για τον συνάδελφο Μόλτερ, να πω στον συνάδελφο Μγκάιερ καταρχά ότι και τον κύριο Ενρίν, τον διευθυντή, τον ενημερώσαμε και τον ε, εκτελεστικό διευθυντή, τον κύριο Φάρκας. Όχι μόνο τηλεφωνικά, αλλά και εγγραφώ έγινε μια ανταλλαγή επιστολών. προκειμένου να μας ειδοποιήσουν, αλλά τότε είχε ήδη συμβεί το κακό. Εκ των υστέρων δεν μπορεί να διορθωθεί αυτό στις, ε, πλευρά, από πλευρά της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού. Υπεύθυνο είναι ένας πάρα πολύ ε, επιμελής υπάλληλο, όποιος θέλει να του ζητήσει αριθμητικά στοιχεία, σίγουρα θα του τα δώσει. Πραγματικά, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορώ παρά να τον υπερασπιστώ τον άνθρωπο αυτό, τον υπάλληλο αυτό. Πάρα πολύ ακριβή και δεν έχω την εντύπωση ότι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χρειάζεται να επισημάνουμε το θέμα αυτό των ε, εξωτερικών υπηρεσιών. Το πρόβλημα είναι γνωστό. Ε, εκατομμύρια δίνουμε για εκμίσθωση κτηρίων. Έμα, ε, είναι δυνατόν να μην χρειάζεται έγκριση. Ποιο το φαντάστηκε αυτό. Με λίγη προσπάθεια θα το είχαμε σκεφτεί, θα το είχαμε φανταστεί. Προσπαθώ να εκφραστώ προσεκτικά. Θα μπορούσαν να το ξέρουν ε, ότι χρειαζόταν έγκριση και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η ίδια η EBA έχει την ευθύνη Με γνωρίζετε σε ό,τι αφορά κτηριακής πολιτικής. Δεν είναι ότι υπάσχω σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ούτε ότι τα μασάω τα λόγια μου. Με σαφήνεια, λοιπόν, το επεσήμενα σε διάφορες περιστάσεις. Άρα δεν μπορώ να σας απαλλάξω από την ευθύνη, δεν μπορώ να σας πω πώς το, εννοεί, εννοούσατε και γιατί συνέβη αυτό που συνέβη. Απλά διαπιστώνω ότι δεν συνέβη αυτό που έπρεπε να συμβεί. Για τον συνάδελφο Μόλτερ, αυτό που είπες σε ό,τι αφορά την ε, γνωμοδότηση αναφέρεται στο σημείο 6 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξαγάγει τα, τα απαραίτητα συμπεράσματα και τις απαραίτητες συνέπειες από το περιστατικό. Τώρα, ποια θα είναι αυτά τα αποτελέσματα και αυτές τις συνέπειες, αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί να είναι δικό μας καθήκον να πούμε ότι κοιτάξτε θα κάνετε αυτό ή το άλλο. Η ίδια η Επιτροπή θα πρέπει να το ελέγξει. Πρόκειται για παραβίαση του κανονισμού για τον προπολογισμό. Οι χρηματοοικονομικές συνέπειες νομίζω και αυτές είναι σαφείς. Η επιθυμία τώρα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και το Ελεκτικό Συνέδριο να ασχοληθούν αυτό το θέμα και αυτό είναι κάτι το σαφές. Καταγγελία των συμβάσεων. Δεν μπορώ αυτό να το απαιτήσω γιατί αυτό θα σήμαινε ακόμα πιο μεγάλο κόστος και θα παρέλειε και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Δεν είναι αυτό ο σκοπός μας. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι στην παρούσα μορφή όπως έχει η γνωμοδότηση περιλαμβάνει όλα όσα μπορούμε να προβάλλουμε ως αξιώσεις, δεν μπορούμε να τα ωρεοποιήσουμε τα πράγματα. Να σας πω ότι στην ΕΣΜΑ τα πράγματα πήγαν διαφορετικά και στην ΕΟΠΑ να σας πω ότι πάλι ήταν διαφορετική η κατάσταση. Και οι άλλε δύο λοιπόν αυτέ οι υπηρεσίε στη Φραγκφούρτη και στο Παρίσι έχουν υψηλέ τιμέ σε ό,τι αφορά την εκμίσθωση των ε, ακινήτων, αλλά τα πήγαν καλύτερα, τουλάχιστον ακολούθησαν τον κανονισμό. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος. Νομίζω ότι αρκετά το συζητήσαμε, το θέμα. Να ψηφίσουμε την όμως που μας την παρουσίασε η Μόνικα εδώ και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ποιο λοιπόν είναι υπέρ της γνωμοδότησης της Μόνικα. Ποιος είναι κατά? Αποχές? Εγκρίνεται. Und wir waren uns, glaube ich, vorher και νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει εξ αρχής ότι σε ό,τι αφορά τα δύο άλλα κτίρια έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θα γνωματοδοτήσουμε και θα τα αφήσουμε τα πράγματα να συνεχιστούν έτσι. Η αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο, η οποία θα πρέπει να έχει ένα ασφαλές κτίριο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Δεν υπάρχει καμία παρανόηση και όλα είναι όπως πρέπει. Δεν θα πρέπει, θεωρώ, να δημιουργήσουμε και επιπλέον δυσκολίες. Είναι φυσιολογικό αυτό. Είναι πραγματικά λογικό αυτό που προτείνεται. Μάλιστα, λοιπόν. Οτιδήποτε δεν μας προβληματίζει, το καλωσορίζουμε. Ωραία. Εντάξει, λέει η Πρόεδρος. Να περάσουμε τότε. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Και να περάσουμε τώρα... Το αγαπημένο θέμα της είναι. σε ό,τι αφορά την προσαρμογή του χρηματοοικονομικού κανονισμού συμφωνία με το MFF. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλι εγώ λυπάμαι. Δεν μπορώ όμως να σας γλιτώσω. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το, το διαπραγματεύσεων το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα αυτά και σε ό,τι αφορά την ευέλικτη διαμόρφωση των μέσων και σε ό,τι αφορά την ε, εγκατάλειψη της ετήσιας αυτής ε, περίοδου και το Connective Euron Facility. Κάναμε κάποιες δηλώσεις το 26 ε, Οκτωβρίου του 2012 και είδαμε λοιπόν ότι ήταν επικοδομητική η στάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υποβάλλει μια πρόταση. Αλλάζουμε μόνο το άρθρο 13 σε ό,τι αφορά την εκπνοή και τη μεταφορά των μέσων. Το C σε ό,τι αφορά τα μέσα για την κατεπίγουσα βοήθεια και στο σημείο D. Το ίδιο και για τα έργα Connecting Europe. Ευέλικτη διαμόρφωση των μη ε, αξιοποιηθέντων μέσων στο σημείο 2, αυτά που αναφέρονται στο πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Εδώ δεν υπάρχει ουσιαστικά προσαρμογή του κανονισμού. Υπάρχουν δύο σημεία στις κοινέ δηλώσει τη 26 Οκτωβρίου 2012 που δεν έχουν εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά το EDF και τον προπολογισμό και τη χρήση των μέσων από την Συμφωνία για τον Καπνό σε ό,τι αφορά δηλαδή το λαθρεμπόριο. Αυτά τα αναφέρω τώρα για να σας ε, παρουσιάσω ποια μέσα έχουμε ακόμα στην ε, τσέπη μας. Να αποφασίσω, θα δω. Ίσως θα σας ε, προτείνω. Δεν ξέρω αν θα κάνω κάποιες καλές τεροπολογίες, Έχουμε ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε ακόμα. Τι θα κάνουμε με την ε, απαλλαγή του PPP για τα joint undertakings. Εδώ είναι κρεμές το σημείο αυτό και γι' αυτό λοιπόν έχουμε μία κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ε, ελέγχου προπολογισμού σε ό,τι αφορά ε, και ζήτησα τη γραμματεία να γίνει μια κοινή συνεδρίαση λοιπόν με την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και να σταματήσει αυτή η διαδικασία και δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπέβαλε συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η δυτή απαλλαγή για το PPP. Έλαβα ένα mail σήμερα από τη Γενική Διεύθυνση και προτείνεται μία ενδιάμεση αναθεώρηση σε ό,τι αφορά την έμεση απαλλαγή. Αυτό δεν είναι αποδεκτό για μας, θα χάναμε την ε, απαλλαγή. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σωστή λοιπόν η στάση της Συγγήτριας σε ό,τι αφορά τις ε, κατεξιοδότηση πράξης του PPP δεν υποβάλαμε αξιώσει σε ό,τι αφορά το PPP αλλά σε άλλα θέματα αναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι, να αναλάβουμε δράση. Θα υποβάλω λοιπόν για το άρθρο 209 ε, μια τροπολογία σε ό,τι αφορά την ε, εκ νέου χρήση των μη αξιοποιηθέντων μέσων. Δεν μπορώ να σας προτείνω κάτι διαφορετικό. Θα τα υποβάλω όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα και θα σας τα δώσω για να τα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ευχαριστώ πολύ. Δύο σχόλια. Καταρχήν, δεν κατάλαβα αν περιμένουμε άλλες τροποποιήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού για την τελευταία συμφωνία γιατί έχουμε τα κίνητρα για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει και αυτά να ενσωματωθούν εδώ. Δεν τα προτείνει η Κομισιόν. Ε, εμείς όμως πρέπει να τα σκεφτούμε εν ώψη της κοινή δήλωσης. Το ερώτημα είναι άλλο. Θες να δρομολογήσεις μια διαδικασία για τις τροπολογίες που θέλει χρόνο. Τώρα, αυτά που αφορούν το πι και αφορούν τη συζήτηση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, αυτό θα ήταν πιο εύκολο να το δρομολογήσουμε ως διαδικασία, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι δυνατόν. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να απαντήσει κατευθείαν ή είναι. Όχι. Ωραία. Έχεις το λόγο λοιπόν. Όχι. Το EDF και τον προπολογισμό του EDF και την ε, συμφωνία για τον καπνό τα αναφέρα σε λεπτομέρειες ε, το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και λέω ότι σε ό,τι αφορά την ε, απαλλαγή δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν θέλω να καθυστερήσω τη διαδικασία. Το θέμα είναι να επιλύσουμε προβλήματα με τον καλύτερο δυνατό πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει να λύσουμε το θέμα της ε, χορήγησης απαλλαγής σε ό,τι αφορά το PPP. Diese andere Geschichte, die du erwähnt hast. Η άλλη ιστορία που αναφέρατε. Δεν την γνωρίζω. Καλό θα ήταν, το συντομότερο δυνατόν βέβαια, να αναλάβουμε δράση. Αλλά στην περίπτωση θα χρειαζόμουν βοήθεια και από σένα. Gibt es den Wunsch der Kommission äh, auf irgend... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει σε κάτι. Ja, bitte. Κύριε Πρόεδρε, ως προς τις συμπράξεις δημοσιοδητικού τομέα, είναι σημαντικό το θέμα. Τα PPP. Δεν καταλαβαίνω. Ομολογώ που πηγαίνουμε και εξηγούμε. Όλοι θεωρώ συμφωνούμε περί του στόχου που είναι η απλούστευση όλος ιδιαίτερος θέλουμε όλοι μας να την απόφαση με τον πιο εύκολο τρόπο για λόγους ε, καλής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η πρότασή μας, η οποία έγινε αποδεκτή από το Κοινοβούλιο, η πρότασή μας λοιπόν στον δημοσιονομικό κανονισμό για τις συμπράξεις ε, αφορά το, 2000, το, το 209, το άρθρο 209, όπου προβλέπεται απαλλαγή μέσω της Κομισιόν. Η απαλλαγή αυτή μέσω της Κομισιόν και το έχουμε εξηγήσει πλιστάκης και νομίζω το δέχονται όλοι με κανένα τρόπο δεν στερεί οτιδήποτε από το δικαίωμα ελέγχου του Κοινοβουλίου. Διότι οι συμπράξεις εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Κομισιόν όσον αφορά την απαλλαγή, αλλά και οι επιχειρήσεις από την άλλη μεριά συνεχίζουν να δουλεύουν πιο εύκολα μέσα σε ένα καθεστώς που εξασφαλίζει δυνατότητες εύκολης διαχείρισης. Πολλές κοινέ ε, επιχειρήσεις αυτό μας είπαν και αυτό επιβεβαιώθηκε και την περασμένη εβδομάδα με την ευκαιρία μιας ε, σύσκεψης που διοργανώσαμε με τη συμμετοχή των εκτελεστικών διευθυντών των ε, γενικών διευθύνσεων και επιχειρήσεων, ιδρυτικών επιχειρήσεων. Και όλοι εξέφρασαν την υποστήριξή του στην αρχική πρόταση της Κομισιόν. 209 λοιπόν, συν κατεξουδότηση πράξη όπως το είχαμε προτείνει. Από εδώ και πέρα τα έχω πραγματικά χαμένα, διότι εμείς προχωρήσαμε για το καλό όλων. Αυτό είχαμε στο μυαλό μας. Και γνωρίζαμε επίσης ότι εάν διαχωρίζαμε, αν αποσπούσαμε τη συμπράξη από την απαλλαγή, τότε τις έξι GTI θα τις ε, θέταμε σε χειρότερη μοίρα από τη σήμερα. και θα είχαμε και πολύ αρνητικέ αντιδράσει από τους ιδιώτες, από τις επιχειρήσεις. Ελπίζω ότι θα έχετε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά. Σήμερα το πρωί μάλιστα υποβάλαμε και πρόταση σύμφωνα με την οποία και το λέω πολύ περιληπτικά ακούσαμε τα επιχειρήματα των επιχειρήσεων και των συμπράξεων και σκεφτήκαμε ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια γενική αναθεώρηση. Και αν δούμε ότι το πράγμα δεν προχωράει, αν θεωρεί δηλαδή το Κοινοβούλιο ότι δεν μπορεί να ελέγξει αυτές τις συμπράξεις, τότε θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε σε μια πιο πολύπλοκη λύση, η οποία όμως θα έκανε πιο δύσκολη τη δουλειά αυτών των επιχειρήσεων. Γι' αυτό λέω και απευθύνω έκκληση σε όλους να κινηθούμε με γνώμονα την απλότητα και την αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό κύριε Κρέσλα. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να καθίσουμε μαζί με το Κοινοβούλιο, να συζητήσουμε ξανά. Ε, υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο και αυτό υποστήριξε την προσέγγιση της Κομισιόν. Και όπως λένε και οι Βρετανοί, ε, χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς ταγκό. Wortmeldungen habe ich jetzt keine mehr. Δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. Α. Εσύ είσαι συγγήτρια. Πάντα θα μιλάς στο τέλος. Ähm, deshalb, also ich gucke mir nochmal um, damit ich hier vergesse. Μην ξεχάσω και κανέναν και ξαναχρειαστεί να το ξανανοίξουμε το θέμα αυτό. Ο Γιένς. Να ζητήσω το λόγο για μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά τα συμπληρωμάτα. Ίσως επειδή να ξεκινήσω από την, από την παρατηρήση. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε το δημοσιονομικό κανονισμό και την οδηγία πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα ταμεία. Υπάρχουν κάποια θέματα που δεν καλύπτονται ακόμα σήμερα. Πότε λοιπόν θα μας υποβάλλετε την πρόταση. Αυτή για τον δημοσιονομικό κανονισμό σε ό,τι αφορά τα joint undertakings τώρα. Μου προκαλεί αρκετά, μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση και έκπληξη το ότι το ακούω αυτό από εσά. Γιατί εγώ και η κυρία Γκρέσλε και με κάποιους υπαλλήλου. Σας επισκεφτήκαμε πριν από κάποιες εβδομάδες και σας ε, όταν φύγαμε είχα την εντύπωση ότι πετύχαμε τον στόχο μας σε ό,τι αφορά την απαλλαγή για τα joint undertakings. Είχαμε μία συνεδρίαση όπου ο κύριος παρατήσει παρουσίασε την απόψή του και έχω την ε, εντύπωση ότι δεν ήταν τελικά αυτά επί των οποίων είχαμε συμφωνήσει την προηγούμενη ημέρα. Είχε ο καθένας φυσικά τα ξεχωριστά του συμφέροντα. Αλλά τώρα νομίζω έχουν περάσει και τέσσερις εβδομάδες και διαπιστώνω ότι βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν και πριν από τη συνάντηση αυτή. Και ένα πράγμα θυμάμαι πολύ καλά από εκείνο το βράδυ, ότι θέλαμε να πετύχουμε έναν διακανονισμό. Έχουν περάσει λοιπόν τώρα τέσσερις εβδομάδες και τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν ε, μου λέτε ότι υπάρχουν νέε καταστάσει και τι να σα πω, μου φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου καινούργια τα στοιχεία αυτά, σαν να έχουμε χάσει τέσσερι εβδομάδε. Και αυτό πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ κρίμα. Ο Γιάννη. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μόνο μία ανταλλαγή απόψεων. Ποια είναι η προθεσμία ε, λήψης απόφασης γιατί όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο μεγαλύτερη ασάφεια υπάρχει. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά μας για να λάβουμε μια τελική απόφαση επί του θέματος. Νομίζω ότι εδώ, Γιάννη, υπάρχουν δύο διαφορετικές προθεσμίες για τα joint undertakings μέχρι τέλη του χρόνου θα πρέπει να έχουμε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Ενώ αυτά που παρουσιάζει είναι, είναι προσθήκες και εδώ δεν υπάρχει κάποιο χρονικό πλαίσιο. Είναι. Για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση θα πρέπει πριν τα τέλη του Ιανουαρίου ε, να τα υποβάλουμε στην Ολομέλεια. Εδώ έχουμε λοιπόν χρονική πίεση, γιατί έχουμε και το θέμα του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου και θέλω να αναφέρω ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα πέρα από το να κοιτάξουμε το άρθρο 209. Κύριε Γενική Διευθυντά, θα ήθελα να σας πω ότι καταλαβαίνω γιατί είσαστε κάπως παρεξηγημένος. σε κάθε αλλαγή και τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού λέμε ότι δεν θέλουμε να χάσουμε κοινοβουλευτικά δικαιώματα. Δεν θέλουμε να τα χάσουμε. Και εδώ θεωρώ ότι έχουμε χάσει ένα δικαίωμα του Κοινοβουλίου. Και αυτό δεδομένων των εξελίξεων και δεδομένων, αν θέλετε, εμ, το, τη σημασία των ε, συμπράξεων στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν μας ε, αρέσει καθόλου προσπαθούμε να τα προσθέσουμε αυτά και σε ό,τι αφορά στα πλαίσια του, της απαλλαγής. Αλλά όλα αυτά βασίζονταν σε μια συνένεση που μπορεί να αφαιρεθεί. Θα μας μείνει λοιπόν το θέμα μόνο του δημοσιονομικού κανονισμού. Σας παρακαλώ να μας καταλάβετε. Είναι το μοναδικό σημείο όπου είπαμε ότι οι πράξεις κατεξουσιοδότηση αποτελούν πρόβλημα για εμάς. Γιατί δεν είναι σαφές και δεν ήταν σαφές ότι με την αλλαγή του τροποποίηση του 209 θα χάναμε τα δικαιώματά μας σε ό,τι αφορά τα joint undertakings. Αυτό ήταν ε, λοιπόν σαφές. Δεν έχω καμία όρεξη να τσακωθώ μαζί σας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρω μία λύση, μία γρήγορη λύση μάλιστα, επειδή σε καμία περίπτωση δεν θέλω να αναστείλω τις διαδικασίες, αλλά δεν έχω καμία άλλη δυνατότητα στην παρούσα φάση. Και η απαλλαγή δεν μπορεί να διανύσετε επαόριστον. Και γι' αυτό λοιπόν είναι στρατηγικό και μόνο το ερώτημα του πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι σε τελική ανάλυση θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την ε, προσέγγιση είναι σαφές, γιατί η Γενική Διεύθυνση Επιστήμης δεν μας αφήνει άλλη δυνατότητα. Και κατά τα άλλα θα ήθελα να υποδείξω ότι είχα και συζητήσεις με τα joint undertakings. Τους ρωτήσαμε ποιον φοβάστε πιο πολύ, εμάς ή την Κομισιόν. Εσάς μας είπαν. Α, μας είπαν όχι ότι σε εμάς θέλουν να μείνουν. Αυτό είναι μια μικρή παρατήρηση. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας δυσκολέψω τη ζωή. Αλλά θα ήθελα να μην αφαιρέσω τη δυνατότητα από το μελλοντικό Κοινοβούλιο να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τα PPP και σε ό,τι αφορά και την αυξανόμενη σημασία του. Αυτό είναι ο μοναδικό λόγο. Θα προσπαθήσω να το προχωρήσω το συντομότερο δυνατόν και να ξαναρχίσουν οι συζητήσει με το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Και γι' αυτό λοιπόν το είπα και έκανα τι σχετικέ δηλώσει, γιατί υπάρχουν ε, κάποια ανοιχτά σημεία από την τελευταία διαπραγμάτευση του δημοσιονομικού κανονισμού Η Συμφωνία για τον Καπνό επιμηκύνθηκε, για παράδειγμα, παρατάθηκε. Αυτό ήταν το σημείο το οποίο ενδεχομένως μπορούμε να το ξαναθέσουμε στο μέλλον και το EDF ρυθμίστηκε στο πολιετές. Δεν θέλω, δεν θέλω να καθυστερήσω τη διαδικασία, ούτε να δημιουργήσω προβλήματα, αλλά την απαλλαγή δεν θέλω να τη χάσω στο σημείο αυτό, γιατί πολύ απλά ε, θα έχουμε πολύ μικρότερη επιρροή σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές αλλαγές. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίρρηση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί αυτό είναι δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε. Ακόμα και αν υπάρχει το παράπονο και η ένσταση ότι αυτό αυξάνει τη γραφειοκρατία. Σε κάποιες περιπτώσεις, το είπα και προηγουμένως, άλλωστε η δημοκρατία έχει το κόστος της το τμήμα της. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Γκρέσλε. Το λέω αυτό όταν παραπονιέται το εκλογικό μου κοινό σε ό,τι αφορά την δημοκρατία. Και ξέρουμε εμείς οι Γερμανοί ότι ποτέ δεν θα γίνει πιο φτηνή η δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Όταν έχει κανείς τέτοιες χιλιετίες δημοκρατίας, μάλιστα. Να περάσουμε στο 7 σημερινή σα διάταξη. Ε, συγγνώμη, το θα το αναβάλουμε. Δεν έχουμε τον εισηγητή μαζί. Εδώ. Και κανένα που μπορεί να αναλάβει τη θέση του για να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Να περάσουμε στο 5. Ο Γιώργος είναι εδώ. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιες αλλαγές οι οποίες πρόκειται να γίνουν. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως υποδηλώνει και το όνομά του Ταμείου Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα από τα μέσα έκφρασης αλληλεγγύης που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου μέσου είναι αντιαφισβήτητη, ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου οι προσπάθειες εξορθολογισμού που καταβάλει πλειονότητα των κρατών μελών καθιστούν την οικονομική ενίσχυση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των καταστροφών ζωτικής σημασίας. Θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θεωρώ ότι στις γενικές γραμμές κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε ένα πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο ταμείο, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της απλοποίησης των κανόνων και των διαδικασιών που του διέπουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί σημαντικά η χρονική διάρκεια μεταξύ του καταστροφικού συμβάντος και της χορήγησης της βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι η ταχύτητα κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης, ενώ και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο στο παρελθόν είχε επικρίνει τη μη έγκαιρη κινητοποίησή του. Επίσης υποστηρίζω την εισαγωγή ενός νέου απλού και ενιαίου ε, κριτηρίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Ελληνικής για τις λεγόμενες έκτακτες περιφερειακές καταστροφές με βάση το δίκτυο του περιφερειακού ΑΕΠ. Θεωρώ ωστόσο ότι το κατώτατο όριο του 1,5% του περιφερειακού ΑΕΠ είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε περιπτώσεις καταστροφών που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις περιφερειακές οικονομίες. Για τον λόγο αυτό προτείνω το το όριο ενεργοποίηση να τεθεί στο 1% του περιφερειακού ΕΠ. Επίση, χαιρετίζω την καθιέρωση τη δυνατότητα να γίνονται προκαταβολέ κατόπιν ετήσεω τη πληγή τη χώρα, το οποίο θα βοηθήσει στην πιο έγκαιρη και άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφών και θα ελαφρύνει την οικονομική επίπτωση στι χώρε, ιδιαίτερα αν αυτέ αντιμετωπίζουν δημοσιονομικού περιορισμού. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω ότι θέτοντα το ανώτατο όριο των προκαταβολών στο 15% του αναμενόμενου ποσού τη οικονομική ενίσχυση, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλά καλύτερα την επιδίωξη για ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση του Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα προκαταβολή, να τονίσω τη λέξη δυνατότητα, κυρία Πρόεδρε, μια και προποθέτει την αίτηση από το κράτο μέλο, δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση αφού το ποσό της προκαταβολής θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό. Ωστόσο θα ήθελα να σας επισημάνω την προσοχή στο ότι η πρόταση της Επιτροπής άρθρο 4α παράγραφος 3 για την χρηματοδότηση των προκαταβολών ως έχει, ως έχει προϋποθέτει αλλαγή του κανονισμού των κοινών διατάξεων το οποίο πριν από λίγο καιρό ψηφίσαμε είναι θεωρώ πολύ προβληματικό και γι' αυτό θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικού τρόπου χρηματοδότησή του. Στη λογική τη όσο το δυνατόν ταχύτερη ενεργοποίηση του Ταμείου Ελληνική κινήθηκε η πρότασή μου. Η Επιτροπή να προβαίνει στην προκαταρκτική αξιολόγηση για το αν μια αίτηση εκπληρώνει τι προποθέσει που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφο 1 τη πρόταση του κανονισμού χωρί καμία καθυστέρηση να υπάρξει ένα ανώτατο όριο πέντε εβδομάδων στον χρόνο που χρειάζεται η Επιτροπή για να αξιολογήσει το κατά πόσο εκπληρώνονται οι προποθέσει κινητοποίηση του Ταμείου και για να καθορίσει το ποσό τη ενδεχόμενη συνεισφορά του. Επιπλέον προτείνω να επεκταθεί το χρονικό διάστημα δυνατότητα χρήση τη ενίσχυση του Ταμείου από 12 στου 18 μήνε για να δοθεί απαραίτητο χρόνο δρομολόγηση των διαδικασιών εκείνων που θα εξασφαλίσουν τη χρηστή διαχείριση των πόρων ιδιαίτερα καθώ η νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων σε πολλέ χώρε είναι αρκετά χρονοβόρα. Άλλο ένα σημαντικό σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η πρόληψη των καταστροφών αποτελεί υψίστη τη σημασίας, καθώς είναι οικονομικώ πιο αποδοτική από ότι η αντιμετώπιση του. Για τον λόγο αυτό το Ταμείο θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Παιδευτικά Ταμεία, ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν συνέργειε με τα συναφή προγράμματα και τους μηχανισμούς που διαθέτει η Ένωση, μεγιστοποιώντας έτσι τον αντίκτυπο της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Σε αυτή την κατεύθυνση επίσης κινείται και η πρότασή μου να καταστεί η τεχνική βοήθεια επιλέξιμη δεπάνη για χρηματοδότηση του Ταμείου Γελεγγύης, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις διοικητικές αρχές των χωρών και των περιφερειών στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί αναγκαίο να μπορέσουν να ενεργήσουν άμεσα και όσο το δυνατόν ταχύτερα σε περίπτωση καταστροφών. Εδώ θα ήθελα να τελειώσω την παρέμβασή μου και αναμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Ähm, José Manuel hat... Σας ευχαριστώ. Το λόγο ζήτησε ο Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria dar os parabéns Ευχαριστώ. Να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί οι προτάσει του στην γνωμοδότηση κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση. Το Ταμείο Αλληλεγγύη, ε, το οποίο υπάρχει από το 2002, ε, έχει χρησιμοποιηθεί σε 23 ε, χώρες και έχουν, έχει αποτελέσει ένα σημαντικό ταμείο για όλα τα κράτη-μέλη. Όλα λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει δυστυχώς έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν το ταμείο αυτό και αυτό νομίζω θα επιδεινωθεί με την αλλαγή του κλίματος. Θα είχα όμως μία ερώτηση να σας κάνω. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής ή κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μου απαντήσει. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι τοπικές καταστροφές να αποτελούν το 1% του ΑΕΠ. Να χρησιμοποιείτε το 1% του ΑΕΠ. Τι γίνεται όμως σε ό,τι αφορά μέχρι τώρα τη χρήση του ταμείου. Υπάρχει κάποια περίπτωση όπου δεν θα μπορούσε να έχει, ε, να έχει χρησιμοποιηθεί το ταμείο εάν ίσχυε δηλαδή ο κανόνας. Δηλαδή, ο νέος κανόνας ε, θα σήμαινε ότι σε κάποια περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσει το ταμείο σε κάποια περίπτωση του παρελθόντος. Δηλαδή, και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η μείωση στο 1%. Αλλά, έχω άλλη μια ερώτηση να κάνω την οποία θέλω να την παρουσιάσω και εν είδη καταληκτικού σχολείου. Υπάρχουν κάποια αριθμητικά στοιχεία τα οποία δεν είναι εύκολα να τα μετρήσουμε σε καταστροφές, για παράδειγμα σε πυρκαγιές. Πρόκειται για μια φυσική καταστροφή. Οι συνέπειες αυτές είναι όχι μόνο προσωρινές αλλά και μακροπρόθεσμες. Πλήττουν μια ολόκληρη περιφέρεια, όλο τον πληθυσμό, το ΑΕΠ, Αυτό όμως ενδεχομένως ε, να μην πλήττεται ε, σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο ε, πανεθνικό ΑΕΠ. Έως τώρα θεωρούσαμε λοιπόν ότι υπάρχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες. Νομίζω όμως ότι σε κάποιες καταστάσεις υπάρχει αυτός αρνητικός μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στο βιωτικό επίπεδο, αλλά αν ορίσουμε τον κανόνα αυτό του 1% ενδεχομένως να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κοινωνικό ταμείο. Και γι' αυτό λοιπόν ε, θα προτείναμε ενδεχομένως κάποια εξαίρεση για τέτοιες περιφερειές. Θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει αυτή η εξαίρεση και στο νέο κανονισμό. Το 1%, το 1,5% θα πρέπει να διευκρινιστεί 1% λοιπόν, όπως προτείνει ο εισηγητής. Θεωρώ ότι είναι καλό ποσοστό αυτό. Κανεί άλλο από πλευρά των συναδέλφων θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σα απαντήσει στι ερωτήσει σα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστώ τον εισηγητή, την γραμματοδότησή του. Ως προς τα ζητήματα που τέθηκαν, έχω τα εξή σχόλια. Η πρόταση να μειωθεί το κατόφλι όσον αφορά το περιφερειακό εισόδημα για να κινητοποιηθεί το ταμείο. Θα για το εξή. Ας πάμε πίσω στην ίδρυση του Ταμείου. Είχαμε στο μυαλό μας τότε πραγματικά μεγάλες καταστροφές. Και έχουμε πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνο όταν είναι δυσανάλογη καταστροφή τότε πρέπει να κινητοποιηθεί η κοινωτική αλληλεγγύη. Σε κανένα σενάριο δεν είχαμε σκοπό να υποκραστήσουμε την εθνική παρέμβαση τους μηχανισμούς που διαθέτει κάθε χώρα. Όχι, επαναλαμβάνω, επρόκειτο, αυτό είχαμε τουλάχιστον στο μυαλό μας, αυτή είναι η συλλογιστική, ε, να αντιμετωπίσουμε πραγματικά εξαιρετικές, σπάνιες, πολύ μεγάλε καταστροφές. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, εάν ταπεινωθεί το κατόφλι αυτό, θα έχουμε περισσότερε δυνατότητε κινητοποίηση του Ταμείου, Βέβαια στο συνολικό ποσό παραμένει το ίδιο. Μάλιστα στο νέο πι τα διαθέσιμα ποσά έχουν σχεδόν καθίσει το μισό. Πώς λοιπόν συγκεράζουμε τις δύο αυτές εξελίξεις. Επαναλαμβάνω, εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο ορισμός της μεγάλης φυσικής καταστροφής. Οπότε προσοχή. Ας είμαστε προσεκτικοί πριν ταπεινωθεί το όριο αυτό κινητοποίησης του Ταμείου. Όσον αφορά το νομικό μέρος, όπως ορθώς ανέφερε ο εισηγητής, η Κομισιόν είχε προτείνει να προσθέσουμε κάποιες διατάξεις στον κανονισμό κοινών διατάξεων για να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Συνοχή και τα διορθωτικά ταμεία. Φτάσαμε στο τέλος της προηγούμενης Προγραμματική περίοδου. Τα πράγματα με τα ταμεία αυτά από εδώ και πέρα γίνονται δύσκολα. Το σίγουρο είναι ότι χρειαζόμαστε ένα κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο θα είναι σαφέ προς όλες τις πλευρές ποιοι είναι οι κανόνες κινητοποίηση του Ταμείου. Όπως είπε και ο Ισίτης, συμφωνώ ότι πρέπει να διευρύνσουμε πρώτα άλλε εναλλακτικέ λύσει αν υπάρχουν βεβαίω. Και τρίτον, όσον αφορά την υστέρηση, το χρονικό περιθώριο εντό του οποίου κινητοποιείται η Κομισιόν. Αν και ο χρόνος που προβλέπουμε ακούγεται παρκή. για ορισμένους η καθυστέρηση αυτή, η υστέρηση αυτή είναι απαράδεκτη. Από την άλλη μεριά, τα αιτήματα υποβάλλονται σε κάποια άλλη γλώσσα ενδεχομένω, χρειάζονται μεταφράσει, θα απεριθούν συμπληρωματικέ πληροφορίε από το κράτος μέλος. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Μετά έχουμε ένα σχέδιο απόφαση τη Κομισιόν, το οποίο και αυτό πρέπει να μεταφραστεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια διάμεσα βήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά. Οπότε ο χρόνος αυτός των ε, πέντε εβδομάδων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πρόχειρη δουλειά ή ανεπαρκή αξιολόγηση των δεδομένων. Κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι τα βασικά μου σχόλια σε αυτή τη φάση. Προτίθεμαι πάντως να συνεργαστώ με τον εισηγητή από εδώ και πέρα και τους βουλευτές για να καταλήξουμε σε συμφωνία επί όλων των σημείων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, θέλεις να... Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και ευχαριστώ τους συναδέλφους βουλευτές για τις προτάσεις τους και τα σχολιά τους. Θέλω ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λήγει στις 17 Δεκεμβρίου. Η προθεσμία για την υποβολή είναι 17 Δεκεμβρίου. Πολύ μόλις πριν τα Χριστούγεννα λέει ο Πρόεδρος. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Κλείνουμε και με αυτό και περνάμε στο σημείο 6. Άλλο ένα αγαπημένο θέμα, κύριε Βέρτμαν, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κύριε Πρόεδρε. Η βάση αυτής της γνωμοδότησης και την ε, καταγωγή της στη μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο από την Κομισιόν όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης του 2014. Μπορώ να συνοψίσω, δυστυχώς, το συμπέρασμα είναι ότι αν συγκρίνουμε το 13 με το 14, συμπεραίνουμε ότι λίγα πράγματα άλλαξαν. Μάλιστα σε πολλούς τομείς δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Λάβατε, θεωρώ, όλες και όλοι το σχέδιο γνωμοδότησης. Εν προκειμένου λάβαμε υπόψη μας την πρωτοβουλία για την επασχόληση των νέων. Ξέρω ότι οι διαπραγματεύσει το ΠΔΠ αποτελούν πλέον παρελθόν. Επισημαίνουμε επίσης το θέμα των ιδίων πόρων. Πρέπει να σχηματιστεί και μια ομάδα για το θέμα αυτό. Υπάρχει περιπτώσει, όπως είπα, υπάρχουν ελάχιστες διαφορές σε σχέση με πέρσι. Το μόνο που έχω να πω με δύο λόγια είναι ότι συνεχίζει να σοβεί βεβαίω η κρίση και θα συνεχίσει να σοβεί. Χρειάζεται πίεση για να πάμε παρακάτω. Ελπίζω ότι θα έχετε σχόλια και παρατηρήσεις τα περιμένω. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 3η Ιανουαρίου. Αν θέλετε να δουλεύετε Χριστουγεννιάτικα, ξεκινήστε να δουλεύετε από σήμερα. Γιατί 22-23 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε εδώ. Η ψηφορία στην ΕΚΟΝ θα προηγηθεί της ένταξης θέματος στην ε, Ολομένια του Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Σχόλια από του συναδέλφου, όχι. Ωραία. Α, συγγνώμη, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Απλώς ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ετήσια έρευνα για το 2014 ε, αφορά και την Κροατία για πρώτη φορά. Εμείς συμμετείχαμε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο άτυπα και για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτίμησε την κατάσταση ε, στις 15 ε, Νοεμβρίου για την διαδικασία αυτή. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι το βασικό ε, χρηματοοικονομικό θέμα που συζητείται στην Κροατία και επίσης ε, συζητείται και ο προπολογισμό του 2014. Συζητήθηκε αυτό το θέμα στο Εθνικό μας ε, Κοινοβούλιο με την Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών η οποία σκιαγράφησε τις ε, βασικές διαδικασίες και αναμένουμε μία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα μας βοηθήσει, θα, ε, θα βοηθήσει να αυξηθεί η ενσυνειδητότητα για αυτό το θέμα, διότι όπως ξέρετε το έλλειμμά μας είναι τόσο υψηλό που η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το θέμα ε, κατά το πρώτο έτος. έτος. Αυτό φαίνεται από τις προβλέψεις, από τις σχετικές προβλέψεις που έχουν ε, ε υποβληθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κανένα άλλο το λόγο. Να σας υπενθυμίσω ότι η 3η Ιανουαρίου είναι όντω η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, αλλά επαναλαμβάνουμε καλύτερο θα ήταν να τα ολοκληρώσουμε όλα αυτά πριν από τα Χριστούγεννα, για να μπορέσουμε με την ησυχία μας να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη κοινή ομάδα εργασίας ε, Επιτροπής ε, Προεδρείου, του Προεδρείου και του ΠΟΥΤΣ, του, του προπολογισμού, δεν συνεδρίασε. Άρα δεν έχουμε κάποια έκθεση σχετικά. Δεν έγινε τίποτα. Μία άσκηση μας δώσανε. Ναι, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Εμείς το δώσαμε αυτό ως άσκηση και το αντιμετωπίζουν στην παρούσα φάση. Μάλιστα. Πολύ λοιπόν συνοπτικά γίνονται αυτές οι εργασίες και αυτοί θέλουν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα λοιπόν. Στο 17. Δεν νομίζω και αυτό να μας πάρει πολύ ώρα. Ο εισηγητής του τριμερούς διαλόγου για την εντολή EIB θα μας μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Εντάχει, Πρόεδρε, βρισκόμαστε στο μέσο της ε, διαδικασίας του τριμερούς ε, διαλόγου. Ε, διαβάσαμε, διατρέξαμε τα κείμενα όλα και τις αιτιολογικές σκέψεις και τώρα συζητούμε με το Συμβούλιο για την διατύπωση των άρθρων και των αιτιολογικών σκέψεων δεν έχουμε ένα σαφές ε, ε, μήνυμα από το, από το Κοινοβούλιο για το επίπεδο δανειοδότησης. Αυτό το θέμα είναι ύψης τη σημασίας, αλλά δεν έχουν συζητηθεί αυτά τα ζητήματα. Περιμένουμε από το Συμβούλιο κάποια γνωμοδότηση εστιάσαμε την προσοχή μας σε κείμενα που άπτονται της διαφάνειας. Εγκρίναμε δύο χρόνια πριν μία ενδιάμεση έκθεση με νέες απαιτήσει για την ΕΤΕ. Χρειάζεται χρόνο όμως, όμως για την ε, εφαρμογή αυτών των προαπαιτήσεων και τώρα υπάρχουν ε, και άλλες απαιτήσει. Θα δούμε τι είναι βιώσιμο και εφικτό γιατί ε, σε ορισμένες προτάσεις είναι δύσκολο να βρούμε έναν ε, ε, ρεαλιστικό τρόπο αντιμετώπισης. Νομίζω όμως ότι αν υπάρχουν διαφορές θα σχετίζονται με, περισσότερο με τον ε, τρόπο ε, ενημέρωσης γιατί το Κοινοβούλιο ε, ζήτησε και εκτεταμένες ε, διαβουλεύσεις με τις επιτόπιες αρχές όταν πρόκειται για πληρωμές και οι οροφές και η περιφερειακή κατανομή, η παρεπόμενη αυτή κατανομή. Έγινε μια τεχνική συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα στον Τριμερή θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε υπό την Προεδρία σας στους ε, τριμερείς. Όλα εξαρτώνται από την απάνταση του Συμβουλίου. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε τελική μορφή πριν από το τέλος του έτους. Θα πρότεινα στους συναδέλφους και στους κοιόδης την επόμενη εβδομάδα να δούμε τα κείμενα τα οποία επεξεργαζόμαστε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες. Νομίζω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουν διευθετηθεί πολλά κείμενα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Γιούτα, θα ήθελα απλώς να επενέσω τον Ιβάιλο, ο οποίος έχει διαχειριστεί τον τριμερή ε, κατά εξαιρετικό τρόπο. Δεν ανήκουμε στην ίδια πολιτική ομάδα, αλλά βρισκόμαστε σε πολύ καλά χέρια. Ναι, σίγουρα. Ο Ιβάιλο λέει ότι εγώ είμαι επικεφαλής του τριμερούς διαλόγου, αλλά αυτό δεν είναι ακριβές. Εγώ απλά είμαι εκεί. Ας το θέσουμε έτσι. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ακριβώς έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να δουλεύουν όσοι πραγματικά είναι ειδικοί, όχι άσχετοι. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη. Ολοκληρώσαμε, με πάση περιπτώσει, ό,τι μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Και θα τα πούμε, λοιπόν, τουλάχιστον στο Στρασβούργο.